So, ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ελπίζω να είχατε ένα θαυμάσιο διάλειμμα για το γεύμα. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Το 9 τη Θεσμική Συμφωνία Πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελβετίας και ανταλλαγή απόψε με τον Κρίστιαν Λέφνα, αναπληρωτή Γενικό Γραμματεία της ΙΕΔ. Πολύ χαιρόμαστε που σας έχουμε και πάλι εδώ μαζί μας. Έχουμε καλέσει και την αντιπροσωπεία συνεργασίας με Ελβετία και Νορβηγία. Να καλωσορίσω και τον Ανδρέα Σουβάμπ, καλώς ήλθατε, που ηγείται αυτής της ε, μόνιμης επιτροπής. Ο κύριος Λέφνα θα μας δώσει κάποια νεότερα στοιχεία σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο με την Ελβετία. Εισαγωγικά εγώ απλώς να πω ότι οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία πλαίσιο δήρυξαν τέσσερα έτη, ολοκληρώθηκαν το Νοέμβριο του 2018, θα θυμάστε ότι είχαμε και στην προηγούμενη θητεία το θέμα αυτό στην ΑΦΕΤ, το Ελβετ Διοικητικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί επί της ε, συμφωνίας αυτής τελεσίδικα. Η Ελβετία είναι ένας από πιο σημαντικού εξωτερικούς εταίρους μα όπω γνωρίζετε με πολύ ε, με αρχαιότατους μάλλον δεσμούς ε, πολιτιστικούς και σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση η συμφωνία αυτή πλαίσιο συνομαδοποιεί τι επιμέρους τομεακέ συμφωνίε που είχαμε με την Ελβετία και υιοθετήθηκε και η σύσταση για, την, για το κείμενο της συμφωνίας αυτής πλαίσιο, με η οποία δίνει, προσφέρει και έναν ε, μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Συνοψίζοντας, θεωρώ ότι η συμφωνία αυτή θα πλαισιώνει, θα συμπληρώνει τις διατάξεις των διμερών μας σχέσεων και διευκολύνει τη συνεργασία με την Ελβετία και σε θέματα εσωτερική αγορά. Θα ακούσουμε τον κύριο Ελέφνα για 10 με 15 λεπτά και μετά θα έχουμε τα ερωτήματα των συναδέλφων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία αυτή να ξαναδούμε το καθεστώς των σχέσεων ευρωπαϊκή Ένωση Ελβετία στα πλαίσια τη συμφωνία Πλαίσιο. Να κάνω ένα βήμα προ τα πίσω για να κάνω μια ιστορική αναδρομή για να σας πω πού βρισκόμαστε και γιατί. Οι σχέσεις αυτές με την Ελβετία έχουν μακρά ιστορία. Η πρώτη άτυπη συμφωνία ήταν το 1972 με τη θέση σε ισχύ της ε, Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών με την Ευετία. Αυτό θα μπορούσε να το θεωρήσει κανείς ε, ενδιαφέρον ιστορικό πλαίσιο, γιατί βεβαίως από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα νομικά και άλλα πλαίσια της συμφωνίας μας, αλλά είναι η πρώτη, όπως σας έλεγα, το πρώτο στάδιο των θεσμικών μας σχέσεων. Διαπραγματευθήκαμε και υιοθετήσαμε μια συμφωνία η οποία περίφθη από τους Ελβετούς πληροφόρους. Ανταυτού αναπτύξαμε την διμερή οδό εντό οικών ώστε να έχουμε μια συνεργασία τομεακή και από τα μέσα προς τέλης δεκαετίας του 90 διαπραγματευθήκαμε μεγάλο αριθμό τομεακών συμφωνιών που καλύπτουν κάθε διάδραση. Άνω των 120 έχουμε αυτή τη στιγμή για διάφορους τομείς δραστηριότητα και για την ελβετική συμμετοχή σε επιλεγμένους ε, τομείς, περιοχές της εσωτερικής αγοράς και του κεκτημένου Σέγγεν. Το ξεχνούμε ίσω, αλλά αρχικά αυτές οι διμερείς τομεακέ συμφωνίες ήταν μια προσωρινή λύση. Γιατί επρόκειτο η Ελβετία να ζητήσει την προσχώρησή της και θα προετοίμαζαν το έδαφος αυτές τις συμφωνίες. Από τότε που δεν είναι επελέχθη πια η οδός αυτή, πήγαμε σε μια σχέση του πολλαπλών συμφωνιών, μιλφέη περίπου λέει ο μιλτής, συμφωνιών, και αρχίσαμε να εξετάζουμε την ύπαρξη ενός πλαισίου που θα μας έδινε μία προβλεψιμότητα και μία συνέπεια στην πλοκή όλων αυτών των συμφωνιών ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε, να εμβαθύνουμε τη σχέση μας να πάμε σε νέε περιοχές και αυτό κατά τρόπον που θα επέτρεπε σε όλους τους φορείς, τους οικονομικούς, τους εμπορικούς, τους πολίτε. να έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη και γνώση του ποιες είναι οι παράμετροι αυτού του πλαισίου κοινών κανόνων. Εξού και η Συμφωνία Πλαίσιο εστιάζεται στην ασφάλεια δικαίου, στην επίλυση διαφορών, στην συνεπή ερμηνεία των κανόνων και των διατάξεων και καθότι μιλούμε και για την εσωτερική αγορά, για την μεταφορά, τη δυναμική μεταφορά του κεκτημένου. Το διαπραγματευτήκαμε αυτό αρκετά χρόνια και καταλήξαμε περί τον ένα χρόνο πριν, δηλαδή ένα, εδώ και ένα χρόνο, καταλήξαμε σε ένα συμπέρασμα το οποίο δυστυχώς δεν έχει επικυρωθεί επισήμω από την ελβετική πλευρά σε μια τιμότητα υπογραφή της συμφωνίας αυτής. Γνωρίζουμε τις ε, προκλήσεις που υπάρχουν, τα προβλήματα που υπάρχουν και τις ε, σεβόμαστε. Παρακολουθούμε την δημόσια διαβούλευση στην Ελβετία που διεξήχθη πέρυσι την Άνοιξη και χαιρετήσαμε και την επιστολή του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, νομίζω ήταν τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, κατά την οποία οι Ελβετοί δήλωναν έτοιμοι να υπογράψουν εφόσον μπορούσε κανείς να λάβει διευκρινήσεις σε τρεις περιοχές. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι ήμασταν έτοιμοι να εργαστούμε επί των διευκρινήσεων που έπρεπε να δοθούν το συντομότερο δυνατόν. Υπάρχει λοιπόν ε, μια διαδικασία εσωτερικής διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και τα ελβετικά καντόνια η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί προτού πάμε στις όποιες διαφημίσεις. Εμείς είμαστε έτοιμοι με πολύ μικρή προειδοποίηση να το κάνουμε αυτό. Και ελπίζουμε ότι θα ολοκληρώσουμε τη συμφωνία αυτή. Η σχέση μας με την Ελβετία είναι πολύ σημαντική. Πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. έχουμε ισχυρές κοινέ αξίες και όραμα, έχουμε σύγκληση πολιτικών σε πάρα πολλές περιοχές, ωστόσο, προκειμένου να προχωρήσουμε στις δυσμερείς μας σχέσεις, πρέπει να έχουμε ένα πλαίσιο κοινών κανόνων, με κοινή ερμηνεία και που θα ισχύουν για αμφότερες τις πλευρές. Και οι κανόνε αυτοί δεν θα πρέπει να καλύπτουν μόνο συγκεκριμένες περιοχές όπως είχαμε τι 120 τομεακές συμφωνίε, αλλά θα είχαμε ένα συνολικό φάσμα για το πλήρες εύρο τη σχέση μας. Στην ουσία δημιουργούμε τις προϋποθέσεις που θα επέτρεπαν στην Ελβετία να συμμετάσχει ευρύτερα σε διάφορα τμήματα ευρωπαϊκής σε ιστορική αγορά, έρευνα, πολλέ περιοχές, πολλά πεδία. Και επομένω. δεν πρέπει να είναι έκπληξη ότι το σημείο κίνηση είναι οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δίκαιο, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και εκεί όπου χρειάζεται η προσαρμογή του υπό τις νομικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να λειτουργεί με τις ιδιαιτερότητες του ελβετικού δικαίου και προκειμένου να προχωρούμε τις σχέσεις μας. Καμιά φορά αφήνεται η εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να επιβάλλει τους κανόνες της εξωτερικό εταίρο Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι παρερμηνία. Δεν προσπαθούν να επιβάλλουμε τίποτα σε κανέναν. Προσπαθούμε να επιτρέψουμε σε ένα στενό εταίρο να συμμετάσχει στην δουλειά μας ή στις περιοχές εκείνες της ιστορικής αγοράς που έχει αποδεχθεί ιδιαίτερα υποφελής για τους οικονομικούς μας φορείς και τους πολίτες. Κατά τρόπον ώστε να μην στρεβλώνεται το πλαίσιο των σχέσεων και της ε, δραστηριότητάς μας. Αυτό επιχειρούμε να κάνουμε με αυτή τη συμφωνία πλαίσιο. Προσαρμόζοντας δηλαδή την εφαρμογή των ευρωπαϊκών διατάξεων προς τις συγκεκριμένες συνθήκες της Ελβετίας. Να σας δώσω ένα-δύο παραδείγματα. Καταρχά, επίλυση διαφορών. Θα έχουμε εδώ έναν μηχανισμό επίλυσης διαφορών και για να καλύψουμε την ανησυχία την ελβετική ότι θα υπήρχε εξωτερική αρμοδιότητα δικαστική αλλά ταυτόχρονα σεβόμενοι και τη βασική μας αρχή ότι τελικός και απόλυτος διαιτητής των κανόνων που διέπουν την εστιατορική αγορά είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εκεί προσπαθούμε λοιπόν μέσω ενός μηχανισμού διαιτησίας να βρούμε μία μέση οδό. Έναν διπλό πυλώνα συνεργασίας για τις κρατικές ενισχύσεις. Κανένας άλλος εταίρος δεν είχε την άδεια να έχει έναν μηχανισμό δύο πυλώνων. Ακόμα και αν δείτε τη συμφωνία απόσυρσης του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν λέγει τίποτα τέτοιο, αλλά στην περίπτωση της Ελβετίας υπάρχει ένα συνταγματικό ζήτημα. μεταξύ δηλαδή ομοσπονδιακού επίπεδου και καντονίων. Καταλήξαμε λοιπόν σε αυτόν τον διτό πυλώνα σχετικά με την εφαρμογή του καθεστώτος των κρατικών ενισχύσεων. Τα συνοδευτικά μέτρα επίσης, τα flanking measures, με σαφήνεια λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες της ελβετικής αγοράς εργασίας. Το περασμένο Μάρτιο, στη σύσταση που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λέγεται ρητά ότι έχουμε μια κοινή ευρύτατη συνεργασία, αμοιβαίω επωφελή επί τη βάση τη κοινή μα ιστορία και των κοινών αξιών. Αυτή είναι μια πολύ καλή περιγραφή, πιστεύω. Αλλά είναι σημαντικό να κατανοεί κανείς και να υπογραμμίζει ότι μέσω της ευρύτατης αυτής εταιρικής σχέσης η Ελβετία έχει πρόσβαση σε υφιστάμενα προγράμματα και δραστηριότητε της εσωτερικής αγοράς. Δεν δημιουργούμε ένα νέο πεδίο που δεν είναι ούτε ενωσιακό ούτε ελβετικό, αλλά ανοίγουμε τις θύρες για την ελβετική πρόσβαση το συμμετοχή σε προγράμματα, σε κοινά προγράμματα. Περιμένουμε με ενδιαφέρον την επικύρωση του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, προκειμένου να προχωρήσουμε αφενός με τις διευκρινήσεις και επί τη βάση των διευκρινήσεων να επιβεβαιώσουμε αυτό που είχε υποθεί στο τέλο τη δημόσια διαβούλευση ότι δηλαδή από πλευράς του θα ήταν έτοιμοι πλέον να υπογράψουν και να επικυρώσουν τη συμφωνία. Και αν μου επιτρέπετε και το σχόλιο, καμιά φορά έχουμε την αίσθηση ότι περιμένουμε τον κοντό, όπως έλεγε και ο Σάμιουελ Μπέκετ. Όσοι το έχετε διαβάσει, η μόνη διαφορά μεταξύ πρώτης και δεύτερης πράξης είναι ότι από το σκηνικό ένα φύλλο από το δέντρο έχει πέσει στο έδαφος. Ένα φύλλο. Τώρα είμαστε λοιπόν στη δεύτερη πράξη. Στο τέλος του έργου οι δύο που περιμένουν τον κοντό λένε πάμε. Και τότε η διεύθυνση του θεάτρου λέει δεν θα συμβεί τίποτα, δεν συμβαίνει τίποτα. Εμείς ελπίζουμε ότι θα συμβεί κάτι. Ότι με αυτές τις διαφημίσεις θα έχουμε ένα επιτυχές αποτέλεσμα προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετίας και όλων μας των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Christian the state of play. Ευχαριστώ, Christian, για την ενημέρωση αυτή. Έχουμε προβλέψει για το σημείο αυτό ε, χρόνο μέχρι τις 3.30 και μετά θα δούμε το σημείο 10 για το Αφγανιστάν. Οπότε έχουμε λίγο χρόνο, απλά πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Βεβαίω θα δώσω πρώτα το λόγο στον ε, πρόεδρο της, της αντιπροσωπείας, τον Ανδρέας Σβάμπ. Ευχαριστώ που μου δώσατε την ε, δυνατότητα να εκπροσωπήσω την αντιπροσωπεία εδώ στην Επιτροπή ΑΦΕΤ και σας ευχαριστώ κύριε Λέφρα και για την εξαιρετικά ολοκληρωμένη παρουσίαση της σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ελβετία. Η αντιπροσωπεία που μόλις την προηγούμενη εβδομάδα συνεδρίασε στο Φαντούτς ε, με τη συμμετοχή και άλλων εταίρων από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ε, ε, έχει τη χαρά να συμμετέχει στη σημερινή συνεδρία τη επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Να σας πω καταρχάς ότι υπήρξαν ε, εκλογές στην Ελβετία ε, που πάντοτε συνοδεύονται από μια κάποια αναταραχή, ξέρετε. Ε, οπότε το ερώτημά μου προς εσάς είναι πώς θα μπορούσαμε με τη νέα Κομισιόν, με επικεφαλή στην Ursula von der Leyen, αλλά και με τα νέα εκλογικά αποτελέσματα που ε, υπήρξαν στην Ελβετία, να επιταχύνουμε τις διαδικασίες ώστε στην ε, Ελβετία να προχωρήσουμε, να οδηγηθούμε σε κύρωση τη συμφωνία αυτή. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε επικοδομητικά να συνδιαμορφώσουμε την ε, διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ λέει ο πρόεδρο, Θα έλεγα επειδή έχουμε χρόνο να απαντάτε σε κάθε ερώτηση αφού θα την έχετε ακούσει και όχι να τι πάρουμε όλε μαζί. Στη συνέχεια έχουμε τους ε, κύριους Μπιουτικόφα και, τον, και Γκάλα. Ευχαριστώ. Σύντομη παρατήρηση για τον κύριο Σβάμπ. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω θερμότατα εσάς προσωπικά και συνολικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την συνεχή στήριξη που μας παρέχετε στη διάρκεια αυτής της ε, διαπραγμάτευσης. Νομίζω ότι η πολιτική αυτή στήριξη και τα ε, ισχυρά πολιτικά μηνύματα ε, μέσω και των ψηφισμάτων που αποσύλλατε ήταν μια πολύτιμη συμβολή στην διαπραγματευτική μας προσπάθεια. Πράγματι, οι εκλογές, οι ευρωεκλογές ε, συνέχεια υπήρξε μια αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έγιναν και εκλογές τον Οκτώβριο στην Ελβετία. Ε, όλα αυτά αποτελούν τομές ε, σε μια συνεχή διαδικασία. Υπάρχει ε, βεβαίως περισσότερη συνέχεια στην πολιτική ηγεσία της Ελβετίας από ότι ε, στην αντίστοιχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και περιμένουμε τον Δεκέμβριο έως ότου συγκροτηθεί σε σώμα το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο μετά τις εκλογές που έγιναν τον Οκτώβριο, για να δούμε και τη σύνθεσή του. Θα ήθελα ωστόσο να συγχαρώ και την ε, απερχόμενη Κομισιόν και τον απερχόμενο πρόεδρο της Κομισιόν, τον Jean-Claude Juncker, ο οποίος προσωπικά επένδυσε πολλά ε, ώστε να προωθηθεί η σχέση αυτή, η διαδικασία αυτή και να θεμελιωθεί σε, γερά, σε γερές βάσεις ε, η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας και νομίζω ότι πρόσφατα σε συνέντευξή του είπε ότι ένα από τα πράγματα για τα οποία μετανιώνει είναι το γεγονός ότι δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, η σύναψη αυτής της συμφωνίας ε, πλαίσιο με την Ελβετία, παρά το γεγονός ότι αυτό, αυτή η αδυναμία δεν οφειλόταν σε έλλειψη προσπάθειας. Η σχέση είναι στέρεη και σταθερή. Βεβαίως μπορεί και να βελτιωθεί και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε με την ε, συμφωνία πλαίσιο. Ελπίζω ότι η νέα ηγεσία της Κομισιόν και το Συμβούλιο θα ε, θελήσει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας με στόχο την ε, όσο το δυνατόν συντομότερη κύρωση της συμφωνίας από πλευράς Ελβετίας. Είπα τον επόμενο μήνα, μόλις ξεκαθαρίσουν τα πράγματα σχετικά με τη σύνθεση του, ομοσπονδιακού, του νέου Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, ε, θα έχουμε πια τη δυνατότητα σε, στο δικό μου επίπεδο αρχικός με τον ομόλογό μου από την Ελβετία και συνέχεια σε επίπεδο Συμβουλίου να ξεκαθαρίσουμε τα ζητήματα που μένουν ακόμη ανοιχτά, να ε, επεξεργαστούμε με κάθε λεπτομέρεια τα θέματα που συμπεριλαμβάνει αυτή η συμφωνία πλαίσια και στη συνέχεια να τα υποβάλουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αντιστοίχω βεβαίω και στο Ελβετικό Κοινοβούλιο προκειμένου να εγκριθούν. Ευχαριστώ. Ο Ράιναρτ Μπιουτικόφα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λέφλερ για την παρουσίασή του. Αν και πρέπει να σας πω, κύριε Λέφλερ, ότι με πολύ ήπιο τρόπο κατά τη γνώμη μου, ε, υιοθετήσατε μια πολύ σκληρή στάση. Συγκρίνοντας, για παράδειγμα, τις διαπραγματεύσεις με την Ελβετία, με το θέατρο του παράλογου. Είναι σαν να υπονοείτε ότι η θέση που υιοθετεί η ελβετική πλευρά είναι παράλογη. Όπως ε, όταν περιμένουμε στο θέατρο τον Κοντό. Νομίζω ότι είναι ε, ιδιαίτερα εταιρική αυτή η προσέγγιση σας ως προς τις διαπραγματεύσεις. Επίσης, ακούγοντάς σας, νομίζω ότι υπάρχει ένας εφημισμός εδώ. Όταν μεταμφιέζεται την πίεση που ασκούμε στην ε, Ελβετία λέγοντας ότι αν έρθουν με το μέρος μας, αν έρθουν με τα νερά μας ε, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε πολλά περισσότερα προγράμματα από όσα τους επιτρέπουμε σήμερα. Ε, αυτό δεν είναι ιδιαίτερα διαφανής τρόπος να επιλύει κανείς υπαρκτά προβλήματα και θα έλεγα επίσης ότι όταν λέτε τα ζητήματα που υπήρχαν ε, έχουν επιληθεί. Ε, πραγματικά δεν ξέρω σε ποια πραγματικότητα ζείτε ή για ποια πραγματικότητα μιλάτε. Κάποιοι από εμά πρόσφατα είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με εκπροσώπους της ε, Ελβετίας από τα συνδικάτα της Ελβετίας και κατά τη γνώμη τους αυτά τα ζητήματα κάθε άλλο παρά έχουν επιληθεί. Και πολλοί από εμά εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο εκφράζουμε ε, τη συμφωνία μας, γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο η προστασία των μισθών και των εργαζομένων. Μιλάμε και για την προστασία του δίκαιου ανταγωνισμού, του θεμητού ανταγωνισμού. Και κάποια από αυτά τα ε, συνοδευτικά ζητήματα, όταν δείτε πώς ακριβώς ε, θα ετίθετο στην πράξη, πολλές φορές οδηγούν σε ανοιχτή παραβίαση ελβετικών κανόνων από εταιρείε που έχουν την, την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ αυτών βεβαίως και γερμανικών εταιρεών. 25-30-35% όλων των παραβιάσεων προέρχονται από αυτές τις εταιρείε. Οπότε νομίζω ότι αιτιολογημένα θα ζητούσε κανείς να επανεξεταστούν αυτά. Τιμώ αυτό που είπα. Σας ευχαριστώ για τις προσπάθειε. Ούτε θέλω να αμφισβητήσω τη συνολική προσέγγισή σα. Ωστόσο, θα ήθελα να παραθέσω τα λόγια του κυρίου Σβάμπ, ο οποίος είπε ότι καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε με μια νέα ορμή τώρα και ενδεχομένως οι περιστάσεις να είναι ευνοϊκές αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται ένα επίπεδο δημιουργικότητας το οποίο θα μπορούσε να μας δώσει τη δυνατότητα να επιλύσουμε ορισμένα πρακτικά προβλήματα χωρίς περιτούς ανταγωνισμούς. Όπως για παράδειγμα όταν προαναγγέλουμε την απόσπαση εργαζομένων διασυνοριακώς. Η Ελβετία, από ό,τι έχω καταλάβει, ε, περιμένουν μια τέτοια προαναγγελία οκτώ ημερών. Με την σύγχρονη τεχνολογία αυτό το πρόβλημα μπορεί εύκολα και με αμοιβαία επωφελή τρόπο να επιληθεί. Εγώ δεν θα επιχειρήσω ότι, ε, να πω ότι ε, μπορούμε πια να οριστικοποιήσουμε τη συμφωνία. Νομίζω ότι πρέπει να επανέλθουμε στα ανοιχτά ζητήματα με ειλικρινή τρόπο για να τα επιλύσουμε. Και σας προειδοποιώ ε, ότι με ένα τέτοιο τρόπο πραγματικά μπορούμε να καταλήξουμε σε, ε, ε σε συμφωνίες αρχές του έτους. Ξέρετε ότι υπάρχει μια πρωτοβουλία πολιτών από την ακροδεξιά στην Ελβετία ξαναλέω για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος από το SVP το οποίο έχει έναν σαφή χαρακτήρα, αντιενωσιακό. Αν δεν λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά τα στοιχεία, τελικά θα διευρύνουμε το χάσμα αντί να το υπερβούμε. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Εντάξει, θα συνεχίσουμε ε, να δίνοντας το λόγο κάθε φορά ε, στον εκπρόσωπο μετά από την ερώτηση, αλλά τρία-τέσσερα λεπτά σας παρακαλώ. Θα ξεκινήσω από το τέλος. Ναι, υπάρχει μια Fox, πρωτοβουλία Fox για επόμε... τον επόμενο μήνα. one ε, ε, ναι, δηλαδή ε, πρωτοβουλία πολιτών. Απ' την άλλη πλευρά ε, λέμε ότι θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η θέση. Μετά θα έχουμε όμως την διαδικασία του Μαΐου και μετά του Οκτωβρίου. Και τι θα γίνει μετά. Ε, αυτό συμβαίνει από το που ζητήσαμε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Εμείς ξεκινήσαμε ε, να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για αυτήν την συμφωνία πλαισίου πριν από δεκαετία. Δεκαετία το τονίζω. Αρχίσαμε τις διαπραγματεύσεις ε, πριν από έξι χρόνια. Δεν είναι δυνατόν να λέει κανείς ότι ε, προχωράμε με μεγάλη ταχύτητα. Είναι το θέατρο του παραλόγου. Όχι. Ωστόσο υπάρχουν κάποια τέτοια στοιχεία παραλόγου. Όταν βλέπουμε ε, να μας λέει ας πούμε την ανάγκη για δημόσια διαβούλευση, να μας τη λέει η κυβέρνηση της ε, χώρας και μετά μας έστειλαν επιστολή και μας είπαν επί τη βάση της ε, διαβούλευσης νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στην διαδικασία, στις διαδικασίες ε, για την, για την επικύρωση μέσα από τρει διευκρινήσει. Αλλά μετά μα είπαν πριν συζητήσουμε για τι διευκρινήσει, θα πρέπει να, ε, κάνει, να γίνουν οι απαραίτητε διαβουλεύσει. Και εμεί είπαμε, μα ε, διαβουλεύσει δεν κάνατε του προηγούμενους έξι μήνε. Εν πάση περιπτώσει, μην ε, ξεχνάτε ότι έχουμε και την περίπτωση του Σάμουελ Μπέκετ και του που περίμενε τον κοντό. Εν πάση περιπτώσει, αναφερθήκατε επίσης ε, στα παρακείμενα μέτρα, flanking measures όσον αφορά την εγγύηση των ε, καταθέσεων, ζητώ συγγνώμη και δεν πρέπει να λέει κανείς, ε, δεν είναι σωστό να λέει κανείς σε έναν βουλευτή ότι κάνει λάθος, αλλά κάνετε λάθος, διότι οι operators στην Ελβετία έχουν αναλογική παρουσία ε, με τους αντίστοιχους ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή αυτοί που δεν ακολουθούν τους κανόνες στην Ελβετία είναι αντίστοιχοι 6-7% των εμπορευομένων. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι σωστό λοιπόν να αναφερόμαστε σε άλλα ποσοστά. Επίσης για τον άλλο κανόνα τον οποίο αναφέρατε. Ε, θα μπορούσε κανείς ε, να στείλει με τέλεξε ή με φάξα παλιότερα τα στοιχεία αυτά. Αλλά τώρα μπορεί κανείς να το κάνει μέσα σε 8 ε, λεπτά. Και συμφωνήσαμε με την Ελβετία ότι οι 8 μέρες, ο κανόνας των 8 ημερών θα έπρεπε να περιοριστεί σε κανόνα 4 ημερών. Μα οι 4 μέρες είναι υπεραρκετές. 80% της εργασίας που γίνεται από τις εταιρείες των ε, ε, εταιρείε ευρωπαϊκέ ε, που στέλνουν αποσπασμένου εργαζόμενους στην Ελβετία ε, χρειάζονται τουλάχιστον πέντε μέρε μέχρι να ολοκληρώσουν τι διαδικασίε για μια απόσπαση που μπορεί να κρατήσει πολύ λιγότερο. Επομένω, ναι, πρέπει να σεβαστούμε ένα σύστημα. Καμία άλλη εταίρο ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει ένα τέτοιο σύστημα. Ο, ο κανόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, μηδενικό. Εδώ προσπαθούμε να προσαρμοστούμε σε ένα άλλο σύστημα. Δίνουμε κάποια λύση δεν είναι εύκολο να το δεχτούν ε, οι χώρες μας στα πλαίσια του Συμβουλίου, αλλά το δέχονται παρόλα αυτά στα πλαίσια μιας ευρύτερης σχέσης. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ο ο κύριος Μπέρκε από την ομάδα ID. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λέφλε, θέλω να σας ε, υποβάλω ένα τεχνικό ερώτημα, γι' αυτό δεν θα μακρηγορήσω. Το 2012 η Γερμανία και η Ελβετία συνήψαν κρατική συμφωνία σχετικά με τις επιπτώσεις του, της λειτουργίας του αεροδρομίου της ε, Ζηρίχης στην επικράτεια της Γερμανίας. Στους τελευταίους 12 μήνες υπήρχαν πολλές διαμάχες και στο κρατήδιο της Βάδης Βιτεμβέργης όσον αφορά την υπέρπτυση, τον θόρυβο που προκαλούν τα αεροπλάνα, τους ε, αεροδιαδρόμους ε, που χρησιμοποιεί το αεροδρόμιο Ζηρίχης. Πιστεύετε ότι αυτή η συμφωνία πλαίσιο μπορεί να επιλύσει ε, αυτά τα εκρεμή ζητήματα που σχετίζονται με την επέκταση του αεροδρομίου Ζηρίχης. Thank Σας ευχαριστώ. Θα είμαι και εγώ ε, σύντομος. Ναι, μα ακριβώς γι' αυτό Προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση για τη συμφωνία πλαίσιο και γι' αυτό θέλουμε να έχουμε ε, έναν απλό μηχανισμό, σαφή και απλό μηχανισμό για την επίλυση διαφορών. Αυτό δεν αλλάζει το περιεχόμενο οποιασδήποτε συμφωνία αερομεταφορών, ε, είτε εσωτερική ή ε, μεταξύ της Ελβετίας και άλλων χωρών ή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας. Όμως από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θέλουμε να έχουμε έναν ισχυρό μηχανισμό επίλυσης διαφορών έτσι ώστε να επιλύονται εύκολα και καθαρά τέτοιου είδους διαφορές. Ο Μιχαήλ Γκάλερ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ σύντομα. Υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις προφανώς εδώ εντός της αιθούσης για τα όσα συμβαίνουν με την Ελβετία. Στην Ελβετία όμως την ίδια με αφορμή και αυτήν την πρωτοβουλία πολιτών, πώς διεξάγεται η συζήτηση. Υπάρχουν διάβλοι για να περάσουμε εμείς τη δική μας ε, θέση, τη δική μας θεώρηση των πραγμάτων, όχι μόνο μέσω της, των επίσημων φορέων, αν θέλετε, των εταίρων μας, δηλαδή ε, στην κυβέρνηση της Ελβετίας, μέσω, ε, για παράδειγμα, εκστρατιών που θα μπορούσαν να, αναλυφθούν. Για μας, βεβαίως, ε, που, εκείνος που έχει την αρμοδιότητα να επιλύει τελεσίδη καταστήματα είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στην Ελβετία όμως είναι τα δημοψηφίσματα. Έχει λοιπόν ε, προταθεί ε, η διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τη συμφωνία. Εμείς μπορούμε ε, με κάποιον τρόπο να περάσουμε το μήνυμα στους Ελβετούς ότι η συμφωνία αυτή υπερασπίζετε και προωθεί και τα δικά σας δικαιώματα ε, γιατί εκεί ε, υπάρχουν πάντοτε προβλήματα και με παραπληροφόρηση. Ε, υπάρχει λοιπόν τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Πολύ καλά γνωρίζετε, λέει ο κύριος Λέφλερ, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 28 χώρες μέλη ε, στις οποίες έχουν ε, οργανωθεί δημοψηφίσματα κατά διαστήματα και για διάφορα θέματα και ξέρετε ε, πόσο ευαίσθητα θέματα είναι αυτά σε εθνικό επίπεδο και γενικώ δεν είναι ιδιαίτερα καλοδεχούμενα από τις εθνικές ας πούμε διοικήσεις. Αυτό γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν κάναμε το ίδιο με μια τρίτη με ένα τρίτο ε, μέρος, με μια τρίτη χώρα που μπορεί να είναι ε, στενή εταίρος, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, αυτό θα μπορούσε να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα και να θεωρηθεί προπαγάνδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεξη στα εσωτερικά κτλ. Αυτό που κάνουμε διαρκώς και συνεχώς είναι μια προσπάθεια εμπλοκής σε δημόσια συζήτηση ε, με παρουσία στα ε, μέσα διαρκώς και σε όλα τα επίπεδα έτσι ώστε να μεταφέρουμε την δικιά μας άποψη ε, για τη σχέση, υπογραμμίζοντας και τονίζοντας τα θετικά στοιχεία της σχέσης και αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο η συμφωνία πλαίσιο μπορεί να προωθήσει ακόμα περισσότερο την σχέση αυτή. Ε, για οτιδήποτε άλλο και οποιαδήποτε άλλη κίνηση θέλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκρουτλέρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Γενική Γραμματέα ε, για αυτές τις ενδιαφέρουσες και πλήρεις ε, επεξηγήσεις. Ο πρόεδρος Γιούνκερ ε, είπε ότι λυπάται πάρα πολύ που στη διάρκεια της θητείας του δεν κατάφερε να ολοκληρώσει αυτό το ζήτημα με την Ελβετία. Μακάρι να ολοκληρωθεί τώρα. Οι σχέσεις ε, με την Ελβετία ε, είναι και παλαιές αλλά και δυνατές, όχι μονάχα σε εμπορικό επίπεδο. Είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πρώτο οικονομικό εταίρο της Ελβετίας, το 52% των προϊόντων που εξάγει η Ελβετία πηγαίνει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, 70% των προϊόντων που εισάγει η Ελβετία εισάγονται, προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως χρειαζόμαστε ε, μια συμφωνία πλαίσιο που ταυτοχρόνως θα σέβεται και τις δύο πλευρές και την Ελβετία και την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε με όλες τις απαραίτητες ε, διευκρινήσεις. Ξέρουμε προστασία των ε, μισθών, των κρατικών επιδοτήσεων, κοινωνικής προστασίας εργασία κλπ. Οπωσδήποτε όμως θα πρέπει να βγούμε από αυτόν τον εκβιασμό κατά κάποιο τρόπο που από την μία πλευρά έχουμε ε, την ε, την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τα χρηματοδοτικά και τα χρηματιστηριακά μάλλον και από την άλλη πλευρά έχουμε ε, την ε, σπάθη των διαφορετικών ταμείων και των χρημάτων του Ταμείου Συνοχής. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η 38η συνεδρίαση της, 20, 7ης και 28ης Νοεμβρίου στο Στρασβούργο έτσι ώστε να είμαστε προάλληλοι active έτσι ώστε οι βουλευτές και από τις δύο πλευρές να προωθήσουν, να σπρώξουν αυτήν την συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Η απάντησή σας κύριε Λέφλερ, ευχαριστώ πολύ. Όπως ε, ήδη είπα, εκτιμούμε ιδιαίτερο στην υποστήριξη που μας έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθ' όλη τη διάρκεια των ε, διαπραγματεύσεων και βεβαίως βασιζόμαστε ε, σε εσά ε, έτσι ώστε να μας δώσετε κίνητρα και να μας οθήσετε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας πλαίσιο και του ανοίγματο που αυτό θα, αυτή θα, θα συνεπάγεται συγγνώμη, για άλλους τομείς. Έχετε δίκιο, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την κοινή συνεδρίαση ε, που θα λάβει χώρα στο τέλος ε, του μήνα, Νοεμβρίου, έτσι ώστε να δούμε ποιες μπορεί να είναι ε, οι προοπτικές. Φαντάζομαι ότι θα έχετε ήδη κάποιες γνωριμίες μεταξύ των Ελβετών μελών, αλλά και θα είναι και κάποιοι νέοι νέα μέλη από πλευράς Ελβετίας. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν να εξηγήσετε προς όλους ε, τις προοπτικές ε, που μπορούν να υπάρξουν μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Δεν νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει ε, να ζητήσει άνοιγμα εκ νέου της διαπραγμάτευσης. Η διαπραγμάτευση ολοκληρώθηκε, έγινε, ολοκληρώθηκε σε επίπεδο Ομοσπονδιακού Συμβουλίου με τον Επίτροπο Χάν. Του του λεχθέντος βεβαίως ε, για να ε, ξαναδοθεί έτσι μία ε, ένταση στην διαδικασία των ε, διευκρινήσεων, ε, νομίζω ότι ναι, μπορούμε ε, να ξαναρχίσουμε τις συζητήσεις και πιστεύω ότι αν καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι θα βρούμε τις απαραίτητες διευκρινήσεις και μετά βέβαια θα ακολουθήσει μια σημαντική εργασία επεξήγησης, παρουσίασης, εκλαϊκισμού κατά κάποιο τρόπο ε, έτσι ώστε να έχουμε την απαραίτητη εμπιστοσύνη και την απαραίτητη στήριξη από τους φορείς ε, ε, και από τις δύο πλευρές. Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ελβετικό Κοινοβούλιο και βεβαίως ως τελικός διαιτητής θα είναι ο λαός της Ελβετίας. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε, μάλλον συνεχίζουμε τώρα Κυρία Σεύκο, ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Λέφνα. Η Ελβετία είναι ο πιο στενό συνεργάτη μα, εταίρο μα. Είχαμε και εισηγητή σχετικά με το θέμα στην προηγούμενη θητεία και μετά πολλά χρόνια διαπραγματεύσεων πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε προδραστικοί ε, ώστε να έχουμε ένα πλαίσιο αμοιβαίως επωφελών ε, συμφωνιών και διατάξεων δεν νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε περαιτέρω αναδιαπραγμάτευση, γιατί γνωρίζουμε που οδηγεί αυτό. Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε κοινή θέση σε αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρετίζει τη συμφωνία αυτή, μέσω της οποίας έχουν πρόσβαση στην ιστορική αγορά οι Ελβετοί και μπορούν επίσης να εκμεταλλεύονται τις τέσσερις βασικές ελευθερίες. Και επομένως Πολύ λυπούμε για αυτά τα flanking measures ε, των Ελβετών ε, και τα πρόσθετα μέτρα ιδιαίτερα για τους εργαζομένους από την Κροατία. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να τονιστεί. Αλλά ε, αναδιαπραγμάτευση τυχόν της συμφωνίας θα άνοιγε το κουτί της Πανδώρας. Για πολλά και διάφορα θέματα που θα μπορούσαν να απελευθερωθούν από το κουτί Πιστεύω λοιπόν ότι δεν θα ήταν καθόλου σοφό να πάμε σε αναδιαπραγμάτευση. Ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Λεφνά. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη. Λέει ο κύριος Λεφνά. Ο κύριος Σικόρσκι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ θαυμάζω την Ελβετία. Είμαι ο παδός της Ελβετίας. Όχι μόνο για τον τρόπο που λειτουργεί η χώρα, Νομίζω ότι είναι πρότυπο πολυ, πολύγλωσσης ομοσπονδίες και δημιουργίας πολυεθνικού αισθήματο πατριωτισμού, λέει ο μιλητής. Τώρα, δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό το ζήτημα καλύπτεται στις διαπραγματεύσεις ή εκαλύφθη, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Εγώ είχα μια εμπειρία εθνικής πολιτικής και μετά ως μέλος εδώ Εκατομμύρια άνθρωποι εκτιμούν, δηλώνουν την ικανοποίησή τους όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει κάτι πρακτικό, επιφέρει μια πρακτική λύση. Ένα από αυτά που ιδιαίτερα εκτιμούν οι νέοι είναι η κατάργηση, λέει ο ομιλητής, του roaming, της περιαγωγής και των σχετικών τελών. Τώρα, στην Ελβετία, μπορεί κανείς να περάσει Χωρί καν να μπει στο έδαφος Ελβετίας, σε διακοπέ για σκι σε ένα βουνό κοντά στα σύνορα και να επιστρέψει σπίτι του και να λάβει έναν εντυπωσιακό λογαριασμό roaming. Εγώ μία φορά έλαβα ένα λογαριασμό 1000 ευρώ για περιαγωγή δεδομένων 24 ωρών. Πρόκειται για κλοπή. Κλοπή λέγω. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Κοιτάξτε, ίσως να μην είναι μόνο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους ε, που επισκέπτονται την Ελβετία. Ίσως να σχετίζεται και με τα Δυτικά Βαλκάνια, λέει ο Πρόεδρος το θέμα αυτό. Εσείς μπορείτε να μας πείτε κάτι. Κύριε Λέφνα. Κοιτάξτε, δεν είμαι ειδικό ε, ε, στις οικονομικές πτυχές των τηλεπικοινωνιών. Το είδαμε το θέμα. Και ε, ναι, υπήρξε ιδιαίτερη πίεση από τους ομολόγους μας να κάνουμε κάτι. Εμείς κοιτάξαμε να δούμε πώς μπορούσαμε εμείς να κάνουμε κάτι. Από ό,τι μου είπαν, στο παρόν πλαίσιο και υπό τις συμφωνίες που έχουμε, θα διακινδυνεύαμε να πάμε σε διαφορά υπό τον ΠΟΕ Δηλαδή άλλε χώρε να μα πούνε «Α, άμα το κάνετε αυτό όμω με του Ελβετούς, το κάνετε και με εμά. Και το οποίο όπω καταλαβαίνετε μα ε, βάζει σε δύσκολη θέση. Είναι ένα μικρό κομμάτι, όχι μεγάλο, αλλά ένα κομμάτι της εξήγηση της πρότασης που υποβάλαμε για τη Συμφωνία Πλαίσιο και τις συνεδεμένες δηλαδή διακηρύξεις δηλώσεις, που αν επικυρωνόταν και ίσχυε, θα εξυγχρονίζαμε τις εμπορικές συμφωνίες με την Ελβετία, ώστε να συμπεριλάβουμε και υπηρεσίες που δεν μπορούσαν καν να εμπίπτουν στο πεδίο της φαντασίας και των ονείρων των συντακτών της Συμφωνίας του 72. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Έχουμε ακόμα πέντε λεπτά προ... πρώτου επομένου θέματος και επομένω η ερώτησή μου είναι η εξή. Φανταστείτε ότι σας περίμενα εδώ απ' έξω ένα κανάλι ελβετικής τηλεόρασης και ζητούσε δήλωση 90 δευτερολέπτων. Το ξαναλέω. Φανταστείτε ότι η ελβετική τηλεόραση εδώ σας περίμενε, εδώ έξω από την αίθουσα, για δήλωση 90 δευτερολέπτων από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση προ του Ελβετού πολίτε που θα πρέπει να κάνω εγώ όταν θα κλείσουμε το θέμα. Εσεί τι θα λέγατε, Έχετε καμιά ιδέα να μου δώσετε. Σε 9 δεύτερα, Πρόεδρε, θα έλεγα just do it, λέει ο μιλητή. ίσως λίγο μακροσκελέστερα θα έλεγα, να εστιαστούμε στην παραγωγική εταιρική μας σχέση και το πώς μπορούμε αυτήν να την προωθήσουμε το συμφέρον των πολιτών μας, λέει ο μιλητής, και των επιχειρήσεών μας, των οικονομικών μας και εμπορικών φορέων. Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να έχουμε ένα πλαίσιο πεδίο κανόνων όπως θέλετε όπου όλοι οι φορείς από τον μεμονωμένο πολίτη μέχρι τις πολυεθνικές θα μπορούν να γνωρίζουν ότι θα την χάνουν ισότιμων κανόνων. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Είναι ένα μικρό κομματάκι από ένα μεγάλο παζλ. Αν λείπει και το παραμικρό κομματάκι από ένα πολύ μεγάλο παζλ, δεν μας φαίνεται έτοιμο το παζλ. Πρόεδρος, ε, ε, συνάδελφοι, δεν ζητήσατε προηγουμένως το λόγο, τώρα λυπούμε, δεν μπορώ πια. Θα συνεχίσουμε σε ακριβώς 60 δεύτερα, ώστε να πάω έξω να κάνω τη δήλωση σε 120 δεύτερα, ώστε να προλάβω να κάνω τη